Uh, uh, Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο σημείο 32 της ημερήσιας διάταξης, εξέταση των τροπολογιών του προγράμματος για τη δικαιοσύνη. Οι εισηγητές είναι ο κύριος Βάιντον Χόλτσερ και η κυρία Χάουταλα. Έχουμε μια κοινή συνεδρία στην Επιτροπή Υποθέσεων και Ελευθεριών του Πολίτη βάσει του άρθρου 35. Τώρα θα ε, καλωσορίσουμε αλλήλους με τον πρόεδρο Μωράη σε αυτή τη συνεδρία. Ευχαριστώ Πάβελ. Όπως είπε και ο Πάβελ, σας καλωσορίζουμε όλους, μέλη της ΛΥΜΠΕ, και ε, αντί του εισηγητού κ. Βάντεν Χόλτσερ θα τον εκπροσωπήσει η κυρία Κάουφμαν. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για την προσέλευση σε αυτή την κοινή συνεδρίαση, όπου προφανώ ε, δύο εισηγητέ θα παρουσιάσουν τι τροπολογίε του. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, οπότε θα δώσω και πάλι το λόγο στον πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σίγουρα θα δώσετε το λόγο τόσο ή άλλο στην κυρία Χάουταλα. Κυρία Χάουταλα, θέλετε το λόγο. Ευχαρίστω, κύριε Συμπρόεδρε. Απλώς να πω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών και των δύο συνεισηγητών ήταν άψογη. Τέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες και τους πιο εισηγητές που συνέβαλαν τα μάλα και με τρόπο πολύ επικοδομητικό στο τελικό αποτέλεσμα στις συμβαστικές δηλαδή τροπολογίες και θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοήθησε να εντοπίσουμε σωστά το πρόγραμμα δικαιοσύνης και το πρόγραμμα αρχών και δικαιωμάτων, αξιών και δικαιωμάτων, για να έχουμε το σωστό διαχωρισμό εφόσον περάσουμε σε τριμμένες διαλόγους και το Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ περισμένες οι διαφωνίες για τη σημασία του προγράμματος δικαιοσύνης. Οι βασικές συζητήσεις που είχαμε επικεντρώθηκαν στο πώς θα λάβουμε υπόψη τις ειδικέ ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Κυρίως πρώτα ποιες ευάλωτες ομάδες θα αναφέρουμε. Δεν μιλάμε απαραίτητο για μειονότητε ή τουλάχιστον όχι μόνον, αλλά κοιτάξαμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και τις πτυχές του, τη διάσταση των φύλων Αναφέραμε τους δικαστικούς λειτουργούς και το δικαστικό κλάδο. Κάποιοι θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ιδιαίτερη στήριξη των ε, δικηγόρων και νομικών που εργάζονται για την κοινωνία των πολιτών. Εγώ θα ήθελα να υποστηριχθεί γενικώ ε, ο κλάδος των δικαστικών λειτουργών. Δεν θα το κάνω τρομερό θέμα για το κείμενο. Αλλά απλώς ε, τονίσαμε λίγο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είχα να πω. Ε, κυρία, η κυρία Κάουφμαν αντικαθιστά τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ. Θέλετε το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολο με μια τόσο εξαιρετική α, εισηγήτρια, την κυρία Χάουταλα και τον εξαιρετικό κύριο Βάιντον Χόλτσερ και οι δύο ουσιαστικά τα ίδια λένε. Και έχουμε λοιπόν δύο επιτροπές, ε, δύο εισηγητές με πολύ μεγάλη εμπειρία και ως η ε, εισηγήτρια της Επιτροπής μου και ως μέλος της ε, Γιούρη και της ΛΥΜΠΕ ότι πραγματικά το κείμενο ήταν πολύ καλό και η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών ήταν πάρα πολύ καλή. Και ίσως όλοι να διαπιστώσατε χθε το βράδυ ότι λάβατε την τελευταία, την τελευταία, τις τελευταίες συμβαστικές πρωτοβουλίες, 29 στον αριθμό, και πολλά θέματα θεωρώ ότι επλήθηκαν πολύ σωστά από κοινού και η κυρία Χάουταλα υπέδειξε ότι ο ορισμός του ποια άτομα θα άμα ωφεληθούν τελικά από τον κανονισμό αυτό. Ήταν πολύ σωστός και καλός σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ε, έχουμε να επισημάνουμε ότι δεν είναι ιδιαίτερη σημασία στα δικαιώματα των παιδιών και φυσικά γίνεται ανάφορα στα θέματα του κράτους δικαίου, μία από τις βασικές αρχές των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών. Και νομίζω ότι στην αξιολόγηση του προγράμματος καταφέραμε να βρούμε και μία λύση η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σε περισσότερο βάθος για το πώς λειτουργήσε το πρόγραμμα και συγκεκριμένα για το ποια άτομα ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα. Άρα θεωρώ ότι συνολικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στέφθηκαν με επιτυχία οι εργασίες μας και να ευχαριστήσω εξ ονόματος του Γιώργου Βάιντεν Χόλτσερ ε, όλους όσους ε, συνεργάστηκαν στην, ε, για την, το κείμενο αυτό. Έχουμε λοιπόν την ψηφοφορία όπως προβλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Σιλβί, λέει ο Πρόεδρος. Και νομίζω ότι το λόγο θέλει άλλος ένας συνάδελφος, ο κύριος Φως και η Καταρίνα. Ναι, σας ευχαριστώ. Εξ ονόματο ε, του σκιωδών εισηγητών από πλευρά του ΕΡΚΑ θα ήθελα να διαβάσω δύο λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δύο εισηγητέ για τη δουλειά που έκαναν έω τώρα και για τι νέε συμβαστικέ τροπολογίε έχουν γίνει σημαντικέ αλλαγέ σε ό,τι αφορά το κείμενο. Αμεροληψία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία των δικαστών είναι ε, όροι και ενίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο και μάλιστα στον διατακτικό. Αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο υποβλήθηκε από πλευρά ε, του ΕΛΚ και χαίρομαι χαιρόμαστε που το έλαβαν υπόψη οι συνεισηγητές. Σε ό,τι αφορά το θέμα του φίλου, εμείς ως ΕΛΚ θελήσαμε να τηρηθεί μια ισορροπία σε ό,τι αφορά το φύλλο και σε ό,τι αφορά την προοπτική για τα παιδιά. Και πιστεύουμε ότι οι νέε συμβαστικέ τροπολογίε λαμβάνουν υπόψη αυτή την προτεραιότητά μα σε ό,τι αφορά την αναφορά τη ε, κοινωνία των πολιτών, στον ορισμό και στου γενικότερου ε, στόχου. Παρά τι κάποιε αλλαγέ, ε, το ΕΛΚΑ ανησυχεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναφορά του κράτους δικαίου και στους ορισμούς και στους στόχους ε, του κειμένου. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα δικαιοσύνης έχει στο επίκεντρο τα, τους επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης, όχι τι ε, των πολιτών και θεωρούμε ότι θα πρέπει να βγει τον ορισμό η αναφορά στην κοινωνία των πολιτών και από τους ε, βασικούς ε, στόχους, αλλά να τηρείται εκεί που αναφερόμαστε σε συγκεκριμένε δράσει και ενέργειε, για παράδειγμα στο παράρτημα του νέου άρθρου 7.1. Σε ό,τι αφορά την καθολική τώρα δικαιοδοσία, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξή, ότι δεν είμαστε αντίθετοι ε, με την αρχή της καθολικής δικαιοδοσίας, γιατί ο σκοπό έχει να καταπολεμήσει την ετοιμορρησία. Ωστόσο, Αναφέροντας τα θέματα καθολικής δικαιοδοσίας, θεωρώ ότι ε, ξεπερνάμε το πεδίο εφαρμογή ε, του κανονισμού και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σε μια τόσο συγκεκριμένη σε ένα τόσο συγκεκριμένο κείμενο. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη τη ε, Κωνσταντινούπολη και την επικύρωση αυτή, αν συμφωνούμε με τη φιλοδοξία των κρατών μελών να επικυρώσουν τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, Μάλλον το, αυτό το μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό δεν συνάδει εδώ, δεν ταιριάζει εδώ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αξιών. Τέλος, ε, θα πρέπει να απλοποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο σαφές ε, το κείμενο, γιατί περιλαμβάνει υπερβολικά πολλές επαναλήψεις σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών. Ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και στην επίτευξη Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνη, οικοδομώντα δικαιοσύνη μεταξύ των επαγγελμάτων στον τομέα τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά και την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω μήπω θέλουν να πάρουν το λόγο οι συγγετές. Η κυρία Κινίτσι πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χάιντερ Βάιντεν Χολτσέρ και την κυρία Χάουταλα. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους, σκιώδεις εισηγητέ, που όλοι συνεισέφεραν στη σύνταξη του κειμένου. Το κείμενο αφορά ένα ζήτημα ζωτική σημασία, την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών σε σχέση με τα μέσα δικαστική συνεργασία και για τι εξελίξει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία στον αστικό και ποινικό κλάδο. Είναι ε, ουσιώδου σημασία για να δώσουμε μια πραγματική και ουσιαστική όθηση στην υλοποίηση του χώρου ελευθερία δικαιωμάτων και ελευθεριών και δικαιοσύνη, στο οποίο νομίζω όλοι προσπογράφουμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η προσπάθεια και ευχαριστώ τους συναδέλφους για το κείμενο που συνέταξαν. Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες μας, ε, ήταν σημαντικό να υπογραμμιστεί η αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων, μια αρχή που ήδη έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βάση της δικαστικής συνεργασίας που βασίζεται στην αμοιβή αναγνώριση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εξίσου σημαντικό, και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους, που δέχτηκαν τις προτροπές μου μέσω των τροπολογιών μου. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε την ε, διεπιστημονική ε, εκπαίδευση των ε, δικαστικών λειτουργών σε σχέση με τα θέματα ανηλίκων. Ήμουν υπεύθυνη για την οδηγία 800 το 2016 για τα ελάχιστα πρότυπα εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών που θα πρέπει να υλοποιηθεί από τα κατημέλη μέχρι τι 11 Ιουνίου τρέχοντο και νομίζω ότι είναι σημαντικό για να διασφαλίσουμε τη σωστή υλοποίηση τη οδηγία αυτή να φροντίσουμε και την εκπαίδευση όλων των δικαστικών λειτουργών που θα κληθούν να την Ταυτόχρονα με τις τροπολογίες μου προσπάθησα να υπογραμμίσω και τη σημασία της εκπαίδευσης των λειτουργών στα σοφρονιστικά ιδρύματα, όχι μόνο στο δικαστικό κλάδο. Για να είναι οι συνθήκες κράτησης αξιοπρεπείς, είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν και εκείνοι ε, που εργάζονται στα ε, σοφρονιστικά ιδρύματα, στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης η κατάσταση εκεί μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Πρέπει να υπάρχει και μια προσπάθεια επανένταξη ε, στην κοινωνία όσων βρίσκονται στη, στα συμφωνιστικά ιδρύματα, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να αντιμετωπιστούν για να αντιμετωπιστούν και οι κίνδυνοι όπω η ριζο, ριζοσπαστικοποίηση, κάτι που είναι ένα πραγματικό κίνδυνο στι φυλακέ και ανησυχεί ω φαινόμενο. Να ολοκληρώσω λοιπόν ευχαριστώντα και πάλι του συναδέλφου για την δουλειά του και στο βαθμό του δυνατού θα συνεχίσω και εγώ να συνεισφέρω στην εξέλιξη του κειμένου μέχρι να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, τους εισηγητές και όσους εργάστηκαν για αυτό το κείμενο. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Κύριε Λεμπρετών, έχετε ζητήσει το λόγο. Κάποιος άλλος, κυρία Ιντβελτ. Και μετά θα επιστρέψουμε στους εισηγητές. Κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα η έκθεση διότι έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αναγκαιότητα την πολιτική ουδετερότητα των δικαστών, εξίσου σημαντικό θέμα και δυστυχώς δεν ισχύει και δεν συμβαίνει σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και οι πιο αρχαίες δημοκρατίες δεν είναι προστατευμένες από αυτή την απουσία, την έλλειψη δυστυχώς πολιτικής ουδετερότητας των δικαστών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπενθυμίσουμε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες. Έχω δύο σχόλια να κάνω. Το πρώτο έχει σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Φως, ε, ο υπενιγμός και η αναφορά στην οικουμενική δικαιοδοσία δεν έχει θέση στο πεδίο εφαρμογής αυτού του κειμένου. Ανοίγει μια, ένα καινούριο κεφάλαιο με τελείως διαφορετική συζήτηση και είναι κακό να τα μπερδεύουμε αυτά. Το δεύτερο σχόλιο μου έχει να κάνει με, με τις ευπαθείς ομάδες και τη βοήθεια. Είναι αδέξιο να ξεκινά κανείς να απαριθμεί διάφορες μειονότητες και να μιλά για την ανάγκη να ανησυχήσουμε για αυτές. Να υιοθετήσουμε άλλη οπτική γωνία και να μιλήσουμε για την ισότητα στην ε, κρίση τη δικαστική, στην ισότητα με τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη μας αντιμετωπίζει. Το να είναι κανείς πολίτης αυτό σημαίνει ότι έχει, υπάρχει ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και πρέπει να έχει συνείδηση αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε πολίτης. Το να επιμένουμε υπερβολικά στις μειονότητες, στο θέμα του φύλου, ενθαρρύνουμε τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας, ακόμα και άθελά μας και διατρέχουμε τον κίνδυνο να ε, οδηγηθούμε σε αυτό τον κοινοτισμό, σε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων εντός της ίδιας κοινωνίας, κάτι το οποίο δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα πουθενά. Δεν θα πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα και δεν θα πρέπει το κείμενό μας να ενθαρρύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Okay. Um, Sophie please. Ευχαριστούμε κυρία Ίντφελτ. Πολύ σύντομα, δεν θα σας ευνηδιάσει ότι διαφωνώ με τον προλαλήσαντα. Συμμερίζομαι πλήρως τα σημεία που έχει προτείνει το ΕΛΚ δεν τα συμμερίζουμε εντελώ μάλλον όλα τα σημεία του ΕΛΚ, αλλά γενικώ η κατεύθυνση που ακολούθησε η συγγήτρια είναι σωστή και σε αντίθεση με το ΕΛΚ χαίρομαι για τις μνήες στην κοινωνία των πολιτών, διότι τελικώς οι πολίτες διοργανώνονται. Είναι σημαντικό να έχουν και αυτοί το λόγο τους και να μπορεί να γίνει ακουστός εδώ. Ευχαριστούμε και τώρα πάλι ο λόγος τους εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις ε, του προσώπου του ΕΛΚ. Ενώ συμφωνώ με την ε, διακρατική ε, δικαιοδοσία, είναι ένας αναδιόμενος χώρος στον τομέα της δικαιοσύνη και κάθε αναδιόμενος χώρος, κάθε κενούργιος χώρος, χρειάζεται εκπαίδευση και χρόνο. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε προσεκτικά τις εξελίξεις Μπορούσε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι εκτός πεδίου του προγράμματος αυτού, αλλά εμένα θα μου φαινόταν περίεργο. Έπειτα, η αναφορά στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι σημαντική γιατί ακόμη και στη δική μου χώρα που θεωρείται ως μία από τις πρωτοπόρους στην ισότητα των φύλων και πολύ αγωνιστική γι' αυτό, ε, παρόλα αυτά έχουμε ένα ε, εμένον πρόβλημα ενδοοικογενειακής βίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορούμε να διαχειριστούμε τις σχετικές υποθέσεις. Και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα μας εξυπηρετήσει. Είναι μια σύμβαση ορόσημο από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξέρω ότι η κύρωση έχει υπάρξει προβληματική ή έχει αποτελέσει ε, αντικείμενο χειραγώγησης από κάποιους που λένε ότι αντίκειται στις οικογενειακές αξίες, στις θεμελίωδες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο κύριος Φως και το ΕΛΚ έχουν δίκιο όταν λένε ότι ίσως υπάρχουν κάποια ζητήματα ως προς τον σωστό διαχωρισμό των δύο προγραμμάτων, της δικαιοσύνης και των αξιών και ε, δικαιωμάτων. Όμως, έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην κατανόηση αυτής, αυτού του διαχωρισμού που πιστεύω ότι μπορούμε να Έχουμε εμπιστοσύνη ότι στα επόμενα βήματα υλοποίηση αυτή τη νομοθεσία θα αποσαφινιστούν πλήρω όλε οι διαφορέ στο, διαχωρισμό των δύο προγραμμάτων. Κύριε Λεμπρετών, ε, σταθήκατε στι ευάλωτε ομάδε και λέτε ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτού, αλλά στι ευάλωτε ομάδε που φτάνουν ενώπιον των δικαστηρίων. Ωστόσο, υπάρχει και το θέμα τη πρόσβαση στα δικαστήρια και ξέρουμε ότι κάποιε ευάλωτε ομάδε έχουν δυσκολία στην πρόσβασή του στη δικαιοσύνη. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Και αυτή θα είναι η πραγματική πράσπιση της ισότητας των πολιτών ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπερβολικό, πολύ ε, υπερβολικά έντονη κοινοτική προσέγγιση. ναι, ε, προσπαθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να οικοδομήσουμε, αλλά ίσως αν εσείς πιστεύετε ότι είναι υπερβολή, ε, σίγουρα βρισκόμαστε σε διαφορετικές οδούς και εμείς θα συνεχίσουμε. Θα ξανασυζητήσουμε πριν ψηφίσουμε στην Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας μέχρι, όπως είπε και η κυρία Κάουφμαν, να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου. Αυτά. Uh, so these were the, the questions from the... Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσει από πλευρά των μελών και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις συμβάσεις και τροπολογίες, τις οποίες θα τις εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας. Για τα θέματα τα οποία δείξατε θα έρθουμε σε επικοινωνία με τον εισηγητή, με τους εισηγητές σε ό,τι αφορά τη διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Προφανώς ε, υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε και αυτό και θα το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι εξαντλήσαμε την ατζέντα της συνεδρίασης αυτής. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα λάβει χώρα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου το απόγευμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ελπίζω να μην έκανε κάποιο λάθος. κάποια στιγμή, προφανώ, κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά θα ελέγξουμε, εν πάση περιπτώσει. Όχι, ελέγξαμε και πραγματικά ε, εκεί θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία. Δεν ήθελα να έχω την τελευταία κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δώσατε την τιμή να συμπροεδρέψω στην ε, συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.